σχετικά με τη δέσμη μέτρων της Επιτροπής για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη και τις Επενδύσεις. Το λόγο λοιπόν έχει ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Γιούνκα. Πρόεδρε, συνάδελφοι, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου κυρίες και κύριοι. Απευθύνομαι, απευθύνθηκα σε εσά πριν από λίγο περισσότερο από ένα μήνα και σας ε, υποσχέθηκα πριν τα Χριστούγεννα να υποβάλω ε, ένα, ε, φιλόδοξο, μια φιλόδοξη δέσμη μέτρων για την ανάπτυξη. Φαίνεται ότι τα Χριστούγεννα έφτασαν νωρί, οπότε είμαι και εγώ εδώ για να υλοποιήσω την υπόσχεσή μου αυτή. Και το κάνω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί εδώ είναι το μέρος που από θεσμικής πλευράς συμβαίνουν τα σημαντικά γεγονότα. Σήμερα η Ευρώπη γυρίζει σελίδα μετά από χρόνια που προσπαθεί να ανακτήσει την δημοσιονομική της ε, αξιοπιστία και να προωθήσει μεταρρυθμίσεις. Σήμερα προσθέτουμε ένα τρίτο σημείο σε αυτό τον ε, κύκλο της εφημερίας με ένα φιλόδοξο ε, πρόγραμμα για την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Η Ευρώπη χρειάζεται ένα τέτοιο πρόγραμμα και η Κομισιόν το παρέχει. Επένδυση στην Ευρώπη σημαίνει κάτι πολύ περισσότερο από ότι νούμερα και χρήμα και λέξεις. Ε, η ανάπτυξη αφορά τους ανθρώπους, τους πολίτες και ιδιαίτερα τους ανέργους. Πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα στους λαούς της Ευρώπης αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Ένα μήνυμα ότι η Ευρώπη επέστρεψε. Δεν είναι στιγμή για να γυρίσουμε να κοιτάξουμε πίσω και να κάνουμε αναδρομές. Οι επενδύσεις έχουν σχέση με το μέλλον. Ασφαλώς θα πρέπει να έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας τις θυσίες των τελευταίων έξι ετών. Δεν θα πρέπει όμως να σταματήσουμε να κοιτάμε το μέλλον, να ανοίξουμε τις αγορές μας και να μεταρρυθμίσουμε αυτά τα οποία δεν λειτουργούν στις οικονομίες μας. Όλα αυτά είναι απαραίτητες συνθήκε, αλλά όχι επαρκή για, την, ε, για την ανάπτυξη. Ασφαλώς και χρειαζόμαστε διαστρωτικέ μεταρρυθμίσει για να εξυγχρονίσουμε και να διατηρήσουμε την κοινωνική οικονομία τη αγορά. Και βέβαια χρειαζόμαστε δημοσιονομική ευθύνη και επιθυνότητα για να ανακτήσουμε την αξιοπιστία μα και να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και για να συμπληρώσουμε αυτό, τον, αυτό το τρίγωνο χρειάζεται ταυτόχρονα και η να ασχοληθούμε με τις επενδύσεις. Και για αυτό το λόγο παρουσιάζουμε αυτή τη δέσμη μέτρων σήμερα. Για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, παρέχει και τα τρία στοιχεία αυτά της επιτυχίας της Ευρώπης για το μέλλον. Μαζί, ε, όχι σε αντίθεση και σε σύγκριση το ένα με το άλλο, αλλά ε, όλα αυτά μαζί σε ένα ενιαίο μήνυμα ότι η Ευρώπη μπορεί να προσφέρει στις επόμενες γενιές και στον υπόλοιπο κόσμο ένα, μια περιοχή η οποία θα είναι ε, ελκυστική για καινούριες θέσεις εργασίας και για επενδύσεις. Γιατί? Γιατί το κάνουμε αυτό. Πρώτον, διότι όχι μόνο έχουμε μείνει πίσω στις επενδύσεις, βρισκόμαστε σε μια παγίδα επενδύσεων, διότι όταν μιλάμε με τους επενδυτές όλοι συμφωνούν ότι η Ευρώπη είναι ελκυστικός τόπος για να επενδύσουν. Αλλά κοιτώντα τα νούμερα, τα νούμερα αναφέρουν, λένε, διηγούνται μια τελείως διαφορετική ιστορία. Οι επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πέσει τα, κάτω από τα 370 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ οι επενδύσεις ε, αυξάνονται στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη έχουν μείνει πίσω. Γιατί, Γιατί οι επενδυτές ε, δεν βλέπουν εμπιστοσύνη, δεν βλέπουν αξιοπιστία. Δεν έχουν εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, διότι αντιμετωπίζουμε ένα σημαντικό παράδοξο. Παρόλη την τεράστια ρευστότητα στις παγκόσμιες αγορές, οι επενδύσεις στην Ευρώπη δεν απογειώνονται. Και τρίτον, διότι οι κρατικοί πόροι ε, για τις χρηματοδοτήσεις έχουν αυξηθεί από το 60% στο 90% σε μερικά χρόνια μόνο. Οι κρατικές δαπάνες αντιπροσωπεύουν αυτή τη στιγμή περίπου το 50% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Χρειαζόμαστε ευφύ χρήση των δημόσιων κονδυλίων ε, έτσι ώστε να ε, ξεμπλοκαριστούν οι ιδιωτικές επενδύσεις. Οι κρατικές επενδύσεις θα πρέπει να κάνουν αυτό που ξέρουν καλά να κάνουν. Χρηματοδότηση των σχολείων, της δημοσιογείας, όχι χρηματοδότηση του ε, χρέους. Σήμερα προσπαθούμε να θεραπεύσουμε αυτές τις ευρωπαϊκές ασθένειες. Ε, έχοντας πάντα στο μυαλό μας την πραγματική οικονομία. Είναι αυτό που πραγματικά είναι σημαντικό. Δεν θέλουμε εθνικές πολιτικές ή ιδεολογικές συγκρούσεις αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε ε, μια συνένεση. Να ξαναγυρίσουμε πίσω στη δουλειά. Ε, ακούγεται ότι χρειάζεται χρειάζεται φρέσκο χρήμα, αλλά εγώ στην πραγματικότητα αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια φρέσκια εκκίνηση, μια καινούρια αρχή εθνικοί προϋπολογισμοί έτσι κι αλλιώς βρίσκονται στο κόκκινο. Ε, η, ε, η ρευστότητα που υπάρχει μας επιτρέπει να μην δημιουργήσουμε καινούργιο χρέος και να λειτουργούμε με ε, ε, προϋπολογισμούς που να μην έχουν ελλείμματα, ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Θα πρέπει να διατηρήσουμε τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για να διατηρήσουμε την αξιοπιστία μας. Όμως, ε, αν τα κράτη-μέλη χρηματοδοτήσουν το ταμείο που προτείνουμε, ε, αυτές οι, οι συσφορές τους δεν θα ληφθούν υπόψη στο Σύμφωνο Σταθερότητας και στους κανόνες του. Θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα καινούριο σύστημα που θα χρησιμοποιήσει τα κρατικά κονδύλια μαζί με μόχλευση ιδιωτικών κονδυλίων που αλλιώς δεν θα μπορούσαν να μοχλευθούν. Κάθε δημόσιο κρατικό ευρώ θα κινητοποιήσει ιδιωτικές επενδύσεις που δεν θα κινητοποιούνται διαφορετικά. Πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά ένα προς ένα τα project. Οι φρέσκες επενδύσεις θα πρέπει να κατευθυνθούν σε σχέδια που να είναι ελκυστικά και που θα δημιουργούν καινούρια οικονομική πραγματικότητα, δεν θα έχουν πολιτικές σκοπιμότητες. Να είμαι σαφής, τα χρήματα τα οποία υποσχόμαστε σήμερα προστίθενται σε αυτά που ήδη υφίστανται. Επιπλέον των 630 δισεκατομμυρίων των διαστροτικών και επενδυτικών ταμείων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Επιπλέον αυτών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Μετά την ε, ε, αύξηση του κεφαλαίου κατά 10 δισεκατομμύρια, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, έχει δεσμεύσει 180 δισεκατομμύρια ευρώ για την πραγματική οικονομία. Και το ταμείο αυτό θα είναι επιπλέον όλων των υπαρχόντων και φυστάμενων προγραμμάτων που ήδη επενδύουν σε υποδομές και ενοτομία και στις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το πιο σημαντικό είναι όμως ότι αυτό το ταμείο ε, είναι ε, επιπλέον αυτών που τα κράτη-μέλη επενδύουν γιατί και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν καλύτερα τα κρατικά κονδύλια και να προβούν σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Να σας εξηγήσω το όραμά μου για το πού πρέπει να πάνε αυτά τα χρήματα. Ε, θυμάμαι τα παιδιά των σχολείων της Θεσσαλονίκης ε, που ε, περπατάνε ε, στι καινούριε τάξει με καινούριου υπολογιστέ. Επίσης ε, έχω στο μυαλό μου καινούρια νοσοκομεία με σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό. Ονειρεύομαι τους γάλους εργαζόμενους να μπορούν να γεμίζουν τις κάρτες τους στα διόδια ηλεκτρονικά ονειρεύομαι ένα ενεργειακό τομέα που θα έχει ενώσει αγορές ε, με, και θα έχει εντάξει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα έχει διαφοροποιήσει τον εφοδιασμό του. Χρειαζόμαστε ε, επενδύσεις ε, που θα αυξήσουν το εμπόριο, που θα ε, μειώσουν τις συμφορίες στους δρόμους. Χρειαζόμαστε πολύ πιο γρήγορο ε, γρήγορα κέντρα διαχείρισης πληροφοριών και ε, πιο ευρυζωνικές ε, επικοινωνίες στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε συστήματα καινοτομίας και έρευνας που αυτή τη στιγμή χρηματοδοτούν πολύ λιγότερο από ότι αυτά των γειτόνων μας και των εταίρων μας. Χρειάζεται να επενδύσουμε περισσότερο στους ανθρώπους. Γι' αυτό μιλάει η κοινωνική οικονομία της αγοράς. Οι ανάγκες είναι τεράστιες. Πρόκειται για το μέλλον των επόμενων γενιών. Πώς θα λειτουργήσει το σύστημα. Τα χρήματα δεν πέφτουν σαν μάνα εξ ουρανού. Δεν έχουμε μηχανήματα να τυπώνουν χρήμα. Θα πρέπει να έλξουμε ε, κονδύλια. Σήμερα δημιουργούμε μια καινούρια αρχιτεκτονική που θα καταστήσει αυτό ακριβώς δυνατό κλειδί είναι να δώσουμε μια ε, δυνατότητα ανάληψης κινδύνου, μια εγγύηση κινδύνου που θα ξεμπλοκάρει πολύ περισσότερες ε, ιδιωτικές επενδύσεις. Τρεις επιλόνες. Πρώτον, δημιουργούμε ένα καινούργιο Ευρωπαϊκό Ταμείο για Στρατηγικές Επενδύσεις που θα ε, εγγυάται με κρατικά κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τον, και τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Το Ταμείο αυτό θα κινητοποιήσει 350 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα τρία χρόνια. Παρ' όλα αυτά κάποιοι λένε ότι ακόμα και αυτό δεν είναι αρκετό. Να σας υπενθυμίσω ότι στην πρόσφατη ευρωπαϊκή ιστορία είναι η μεγαλύτερη προσπάθεια που έχει γίνει ποτέ σε ε, κονδύλια τα οποία θα δημιουργήσουν καινούριε επενδύσεις χωρίς να αλλάζουμε τους κανόνες. Γνωρίζω ότι ορισμένοι από εσά ανησυχούν για, για τα κονδύλια, για την έρευνα και τις υποδομές. Ε, φοβούνται ότι θα αφαιρέσουμε χρήματα από τον ορίζοντα 2020 ε, και ε, ότι ποσά θα χαθούν. Όχι, δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. το αντίθετο θα συμβεί. Δεν μετακινούμε χρήματα από τη μία γραμμή στη μία, σε μία άλλη, βελτιώνουμε και μεγιστοποιούμε την απόδοσή τους. Αν τα κράτη-μέλη επίσης συνεισφέρουν στο Ταμείο, τότε το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ακόμα υψηλότερο. Αξιότιμοι κυρίε και κύριοι, το δεύτερο στοιχείο, δεύτερο άξονα του προγράμματό μα είναι ο εξή. Ε, θα έχουμε μία αξιόπιστη γραμμή επενδύσεων που θα στηρίζεται από επενδύσεις ε, οι οποίες ε, θα στηρίζουν προγράμματα που και αυτά με την πλευρά τους βοηθούν την ανάπτυξη. Δεν είναι η δουλειά των πολιτικών να εκτελούν προγράμματα. Θα έπρεπε να είμαστε λιγάκι πιο μετριόφρονες. Αυτό είναι το καθήκον των εμπειρογνωμόνων οι οποίοι διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία όπως επίσης και την εμπειρία για να πράξουν κάτι τέτοιο. Το Ταμείο λοιπόν θα στηρίζεται από μια ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η οποία Επιτροπή θα επιλαμβάνεται και θα αξιολογεί κάθε πρόγραμμα το οποίο θα υποβάλλεται και το οποίο θα πρέπει να προσφέρει υπεραξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τρίτο στοιχείο, ο τρίτος άξονας του προγραμματός μας είναι ένας πολύ φιλόδοξος χάρτης πορείας με τον οποίο επιθυμούμε να καταστήσουμε την Ευρώπη πιο ελκυστική. Είναι Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, είναι καθοριστική σημασία και για το λόγο αυτό θα θελήσουμε να άρουμε τις ε, κανονιστικές περιοριστικές ρυθμίσεις. Γιατί δεν πρόκειται μόνο για το οικονομικό επίπεδο, το δημοσιονομικό, πρόκειται κυρίως για τις σωστές συνθήκες πλαίσιο σε κανονιστικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων τα τελευταία χρόνια εργάστηκε αποτελεσματικά και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για το γεγονός ότι μπορώ να την έχω ως εταίρο σε αυτή την προσπάθειά μου του επενδυτικού προγράμματος. Το 3α της ε, τράπεζας που βεβαίως και αυτό δεν σημαίνει ότι εξαιρείται από οποιοδήποτε κίνδυνο. Αυτό αποτελεί ένα ατού το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα για την Ευρώπη. Χωρίς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν θα μπορούσαμε να έχουμε φτάσει στο εν, λόγω πρόγραμμα επενδύσεων και θα ήθελα να ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζα Επενδύσεων, τον κύριο Χόια, με τον οποίο είχαμε τα τελευταία χρόνια μια ιδιαίτερα αγαστή συνεργασία. Επιτροπή, γνωρίζετε, ε, έχει αναλάβει τα καθήκοντά της μόλις τους ε, τελευταίους τρεις μήνες, αλλά ο κύριος Βέρνα Χόια ήδη κατά τον Ιουλίο, πριν αναλάβω εγώ τα καθήκοντά μου, ε, συνεργαστήκαμε και οφείλω να ομολογήσω ότι του είμαι ευγνώμων και επίσης και ιδιαίτερα ευτυχής ε, και για το γεγονός ότι με την άδεια του Προέδρου του Κοινοβουλίου μπορεί να παρίσταται σε αυτή τη συνεδρίαση. Κυρίες και κύριοι, έχουμε μπροστά μας σημαντικά βήματα που πρέπει να κάνουμε γιατί βρισκόμαστε μόνο στην αρχή. Για το λόγο αυτό επιτρέψτε μου να απευθυνθώ σήμερα σε όλους οι οποίοι επιθυμούν να επανέλθει η Ευρώπη σε ισχυρή ανάπτυξη τα κράτη-μέλη πρέπει να ενταχθούν στο Ταμείο και με τον τρόπο αυτό να στηρίξουν περαιτέρω την αποτελεσματικότητα του Ταμείου. Γιατί και τα κράτη-μέλη οφείλουν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους οποτεδήποτε πρόκειται για την ανάκαμψη στον τομέα των επενδύσεων. Οποιοδήποτε ευρώ δαπανάται από τον κρατικό κορβανά μπορεί να αποφέρει 15 ευρώ. Ανταυτού εγώ σας υπόσχομαι ότι αυτές οι κεφαλογικές συνεισφορές στο Ταμείο θα ληφθούν υπόψη κατά την επανεξέταση των ε, προπολογισμών όμως δεν θα είναι εις του προγράμματος ε, σταθερότητας. Ε, διερωτάται κανείς γιατί να πρέπει τα κράτη-μέλη να συνεισφέρουν εάν δεν μπορούν ευθύς εξ αρχής να γνωρίζουν τι θα αποκομίσουν για την ίδια τους τη χώρα. Είναι πάρα πολύ απλό. Κοιτάξτε, η μεγαλύτερη ανάπτυξη στη Γαλλία είναι εξίσου καλή και για ανάπτυξη στη Γαλλία. Το ίδιο ισχύει και για τη Γαλλία. Μεγαλύτερη ανάπτυξη στη Γαλλία σημαίνει μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ιταλία στη Νότια Ευρώπη. Αν υπάρξει ανάπτυξη, αυτό θα είναι καλό για τη Γερμανία. Επιτέλους, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε μια κοινωνία που μας συνδέει, μια κοινή μοίρα, μια κοινότητα με ευθύνες και υποχρώσεις. Όσον αφορά λοιπόν τα 315 ε, δις ευρώ που είναι ο στόχος μας δεν πρόκειται για ανώτατο όριο. Γιατί αν το Ταμείο εντωμεταξύ αποδειχθεί αποτελεσματικό που θα συμβεί κάτι τέτοιο και είμαι σίγουρος θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το ποσό τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο νομίζω ότι θα έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη αυτού του επενδυτικού προγράμματος. Αυτό που χρειαζόμαστε στην Ευρώπη είναι ένα ένας ε, συνασπισμός των προθήμων για επενδύσεις. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πραγματικά βασίζομαι στην δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να εγκρίνουμε τη σχετική νομοθεσία το γρηγορότερο δυνατό προκειμένου να θεσπιστεί το νέο αυτοταμείο. Και καλό λοιπόν και του συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να πράξουν αναλόγω. Θα πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί το Ταμείο αυτό μέχρι τον Ιούνιο του 2015, προκειμένου να είμαστε πραγματικά σε θέση να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πάρα πολύ σημαντικός εταίρος, προκειμένου η Ευρώπη να καταφέρει να κάμψει οικονομικά. Εμεί, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούμε ότι είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σα και οι εκπρόσωποι του νέου αυτού ταμείου θα πρέπει να έρχονται πολύ συχνά εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να σας λένε ακριβώς τι πράττουν. Θεωρώ λοιπόν ότι ε, όλοι οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς επίσης και οι εκπρόσωποι του ταμείου αυτού, αλλά και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, θα πρέπει πολύ συχνά να υποβάλουν εκθέσεις συγκεκριμένες εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παράλληλα όμως θα πρέπει να είμαι απόλυτα σαφής. Έχουμε την απόλυτη ανάγκη της δικής σας έγκρισης και της δικής σας υποστήριξης. Σε καμία περίπτωση θα πρέπει να πολιτικοποιηθεί το Ταμείο αυτό. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να παίξουμε κάποιο πολιτικό παιχνίδι σε σχέση με το Ταμείο αυτό. Δεν πρέπει να παίξουμε κάποιο εθνικό πολιτικό παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να ελοποιήσουμε το Ταμείο αυτό προκειμένου να πείσουμε τους ιδιώτες ε, επενδυτές και τις αγορές. Και βασίζομαι προφανώς στον επαγγελματισμό, την εμπειρία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προκειμένου να γίνει κάτι τέτοιο. Το σχέδιο λοιπόν αυτό δεν θα πρόκειται σε καμία περίπτωση να αποτελέσει μία τράπεζα η οποία θα δίνει χρήματα με έναν τρόπο πάρα πολύ περιοριστικό ή απόλυτο. Αντίθετα, χρειαζόμαστε την απαραίτητη ευελιξία στα πλαίσια αυτού του μηχανισμού. Ένα μηχανισμό ο οποίος θα μπορεί πραγματικά να προσαρμόζεται στις νέες ανάγκες. Ένας μηχανισμός ο οποίος ε, δεν θα προβλέπει θεματικά τομεακά στεγανά όπως είχαμε στο παρελθόν. Χρειαζόμαστε έναν αξιόπιστο νέο μηχανισμό, ο οποίος θα είναι σε θέση να εγγυηθεί ένα υψηλό επίπεδο ευθύνης. Έναν μηχανισμό ο οποίος ήταν σε θέση να υποστηρίξει περισσότερο τις χώρες εκείνες οι οποίες επλήγησαν ιδιαίτερα από την κρίση, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες επενδύσεις σε αυτές τις χώρες. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να οργανωθούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι λοιπόν, ένα μήνα μετά την θέση σε ισχύ τη Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναλαμβάνουμε τι ευθύνε μα και σα κάνουμε μια συγκεκριμένη πρόταση. Καλούμε και εσά όμω να λάβετε τι ευθύνε σα, καλούμε και εσά να διαδραματίσετε τον δικό σα σημαντικό ρόλο. Ήδη από σήμερα σα λέω ότι αν το σχέδιο αυτό λειτουργήσει και είμαι πεπισμένο ότι θα λειτουργήσει, τότε θα συνεχιστεί και για το 2018, 2019 και για το 2020. Κύριε Πρόεδρε, Πρόκειται λοιπόν για μια επένδυση που κάνουμε αυτή τη στιγμή προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε την οικονομική μας πολιτική. Επικεντρωνόμαστε στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μακροπρόθεσμες θέσεις απασχόλησης. Θέλουμε να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες πραγματικά μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης και μπορούν να συμβάλλουν στο να ανακάμψουμε οικονομικά. Κυρίες και κύριοι, κάνουμε αυτή τη στιγμή μια έκκληση όσον αφορά την δημοσιονομική ευθύνη, όσον αφορά νέα επενδυτικά όργανα, νέα επενδυτικά σχέδια, προκειμένου να λειτουργήσει το νέο αυτό σχέδιο, να λειτουργήσει το νέο αυτό ταμείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να εμπλέξουμε περισσότερο και τις κυβερνήσεις. Θα πρέπει να βασιστούμε λοιπόν σε τρει τομεί. Σχέδια, χρηματοδότηση και τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να δημιουργηθεί ένα θετικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Κατά αυτόν τον τρόπο εμφυσούμε νέα ελπίδα σε εκατομμύρια Ευρωπαίων οι οποίοι έχουν απογοητευθεί από όλα αυτά τα χρόνια τη κρίση. Όντω η Ευρώπη, το πιστεύω, μπορεί να αποτελέσει επίκεντρο σημαντικών επενδύσεων. Ναι, η Ευρώπη μπορεί να προχωρήσει μπροστά και ναι, το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο θα επιζήσει. Αυτή τη στιγμή κινούμαστε λοιπόν στην ε, σωστή κατεύθυνση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να επιστρέψουμε πίσω. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιούγκα. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων το λόγο έχει ο κύριος Χόια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και κυρίω, σας ευχαριστώ πολύ για το γεγονός ότι μου κάνετε σήμερα την τιμή να μπορώ να παρίσταμαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επίση να σχολιάσω το πρόγραμμα που έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, θα ήθελα λοιπόν να προτείνω στην τράπεζα να στηρίξει το πρόγραμμα που παρουσίασε μόλις πριν από λίγο ο κύριος Γιούνκα και να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις ε, που αφορούν στη δουλειά της τράπεζας κατά τους επόμενους μήνες. Ε, βεβαίως το Δεκέμβρη θα κατετεθούν οι προτάσεις στο αρμόδιο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών και στο Συμβούλιο Κορυφής το Δεκέμβρη. Θέλω να σας πω ότι είμαστε ακράδαντα πεπισμένοι ότι πρέπει να προχωρήσουμε στο θέμα των επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις αρχές του έτους η Τράπεζα εκπώνησε μία μελέτη σχετικά με το επενδυτικό χάσμα που υπάρχει στην Ευρώπη. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι πλέον για 7 συναπτά έτη η Ευρώπη είναι κάτω από τα στοιχεία του 2007 κατά τουλάχιστον 20% και αυτή η τάση εξακολουθεί να υπάρχει. Πέρα από αυτό, για περίπου 15 συναπτά παλιέτη, εμείς βρισκόμαστε σε χειρότερη θέση ε, σε ισχυρότερη σχέση με τους ανταγωνιστές μας, οι οποίοι δεν βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εκτός αυτής. Και σε σύγκριση με κάποιους από τους ε, περισσότερους πιο αναπτυγμένους από αυτούς είμαστε και κατά περίπου 1% του ΑΕΠ κάτω από τις επενδύσεις που επενδύουν εκείνοι για την έρευνα και την τεχνολογία. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να λάβουμε μέτρα. Προτείνω λοιπόν ή θα προτείνω στο ΕΚΟΦΗΝ καταρχήν να εκπονηθεί μια μελέτη για να διαπιστωθεί κατά πόσον ο ισχυρισμός ότι δεν υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες, κατά πόσον αυτό ευσταθεί ή όχι. Ε, έγινε ήδη μια μελέτη η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μόνο ημέρες και ε, κατέδειξε ότι παρότι ενδεχομένως υπάρχουν κάποιοι ευκταίοι πόθοι, ε, υπάρχουν προγράμματα, υπάρχουν ιδέες και απόψεις και πρέπει να υπάρχουν. Παραμένει λοιπόν το ερώτημα το γιατί δεν καλύπτεται αυτό το επενδυτικό κενό από τον ιδιωτικό τομέα και από όλου του άλλου που μπορούν να συμβάλλουν. Ποια είναι τα εμπόδια ω προ τι επενδύσει, ενδεχομένω στην πλευρά των κινητήρων, μα αν είναι πρέπει να του αντιμετωπίσουμε στον κανονιστικό τομέα, στον νομοθετικό τομέα. Με μεγάλη μου χαρά άκουσα τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που λέει ότι είναι αποφασισμένο να επιληφθεί και αυτών των θεμάτων. Υπάρχει βέβαια και το θέμα τη εμπιστοσύνη που είναι καθριστική σημασία για όποιον οποιοδήποτε, για οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση ληφθεί στο μέλλον. Άρα δηλαδή τα πράγματα πρέπει να τα έχουμε σε μια αλληλουχία. Καταρχήν, εντοπισμό του επενδυτικού χάσματο. Δεύτερον, τα αίτια, γιατί δεν καλύπτεται το κενό. Και τρίτον, τι θα κάνουμε σε σχέση με όλα αυτά. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή τα τελευταία 7 χρόνια της κρίσης. Από το 2007 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα διέθεσε πάνω από 500 δις για επενδύσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και μέχρι του χρόνου θα έχουμε ε, διαθέσει 108 επιπρόσθετα δις για επενδύσεις, ε, κάτι που πρότεινε το ε, Συμβούλιο Κορυφής ε, του 2012. Τότε δεν ήμουν σίγουρος ότι θα μπορούσαμε κατά 18 φορές να αυξήσουμε το ποσό, αλλά θέλω να σας πω το εξής, ότι φαντάζομαι του χρόνου που θα έρθω να σας ξαναβρω θα έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ αυτά τα 108 δις που σκοπεύουμε να διαθέσουμε για την Ευρώπη. Πριν λοιπόν από την κρίση τα προγράμματα χρηματοδοτούνταν άμεσα από το δημόσιο τομέα, ο οποίος αναλάμβανε κυρίως τον κίνδυνο. Οι δημόσιες δαπάνες για τέτοιου είδους προγράμματα τώρα έχουν μειωθεί, βρισκόμαστε σε υποεπενδυτικό κλίμα και αυτό αποτελεί κίνδυνο για τις οικονομίες μας. Όμως σε σχέση με τις ζωφερές ημέρες τώρα πλέον η ρευστότητα υπάρχει και μπορούν να διατεθούν κονδύλια για τα ασφαλέστερα των προγραμμάτων. Βεβαίως ε, υπάρχουν ε, κάποιες, κάποιες ενδείξεις στην αγορά που βοηθούν στο να αντιμετωπίζονται κίνδυνοι και εξακολουθούν όμως να υπάρχουν κάποιες ανησυχίες. Εδώ θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει όμως μια ε, μαγική συνταγή γιατί η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ρευστότητα είναι κάτι που ποικίλει στα κράτη-μέλη και πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με πολυσχηδή και διαφορετικό τρόπο. Είναι λοιπόν σημαντικό να αντιμετωπίσουμε Τη τις αποτυχίες αγοράς που εξακολουθούν να αποτελούν κίνδυνο για τις επενδύσεις. Αυτά θα ενταχθούν στο επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο όπως σας είπα θα εξεταστεί στο πλαίσιο του ταμείου που πρότεινε ο Πρόεδρος. Θα προτείνω στο ΕΚΟΦΗΝ και στο Συμβούλιο Κορυφής η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να συμβάλλει με 5 δις ευρώ σε αυτή τη νέα πρωτοβουλία. Άρα θα μιλάμε για 16 δις ευρώ από τον κοινοτικό προπολογισμό, κάτι που εκκρεμεί ακόμα να επιβεβαιωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς θα μπορέσουμε να αυξήσουμε τα προγράμματα ε, σε σχέση πάντα με την αξιολόγηση του κινδύνου και θεωρούμε ότι το 2015 θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την ήδη υπάρχουσα υποδομή. Και αυτό είναι το πλονέκτημα. Είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να λάβετε σημαντικέ αποφάσει. και το Συμβούλιο επίση θα κληθεί να το πράξει αυτό. Άρα θα χρειαστεί κάποιο χρόνο μέχρι να υπάρξουν αυτέ οι νέε υποδομέ. Εμείς είμαστε σε θέση να καλύψουμε αυτό το χρονικό κενό έτσι ώστε ήδη από τι αρχέ του 2015 να υπάρχουν σημεία επιτυχία. Με απλά λόγια. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ένας σημαντικός ε, χώρος, μια σημαντική πηγή. Εμείς αναπτύσσουμε δραστηριότητες και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατόπιν τούτου θεωρώ ότι είμαστε ένας απαραίτητος εταίρος που στηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε όλες τις πολιτικές, τις ανθρωπιστικές, ε, τις κλιματικές και άλλες. Θεωρούμε ότι οι προτινόμενες πρωτοβουλίες πραγματικά θα οδηγήσουν στο να ξεκλειδώσουν οι πραγματικέ επενδύσεις στην Ευρώπη. Ευρωπαϊκή Τράπεζα γνωρίζει ότι αυτό δεν είναι ένα είδος ε, μαγικής λύσης, αλλά είναι η δική μας η συνεισφορά ε, που θα καταδείξει για άλλη μια φορά ότι εμείς είμαστε εκείνοι που μπορούμε να κάνουμε διαφορά. Και το ξέρουμε αυτό κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Vielen Dank, Herr Heuer. Wir kommen jetzt zur Das Wort hat für die Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χόια. Το λόγο λοιπόν έχει τώρα εκ μέρους του ΕΛΚ ο πρόεδρος του, ο κύριος Βίμπερ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Χόια, αξιότιμοι συνάδελφοι, ε, Υποσχέθηκα στον κύριο Γιούγκελ όταν εξελέγει και κατά τη διάρκεια τη προεκλογική ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το επίκεντρο θα είναι οι πολίτε. Γι' αυτό λοιπόν ε, υπογραμμίζω και υποστηρίζω ανεπιφύλακτα αυτά που είπε ο κύριο Γιούγκελ ότι μιλάμε για του άνεργου, μιλάμε για τι επιχειρήσει που θέλουν να επενδύσουν, μιλάμε απλά και μόνο για τον άνθρωπο, για πρακτικά προβλήματα. Θα ήθελα λοιπόν να αποτίσω φόρο τιμή στην Επιτροπή για το γεγονό ότι μέσα σε τρει και μόνο εβδομάδε καταθέτει αυτή τη δέσμη μέτρων την επενδυτική. Επίσης δείχνει ότι είναι ενωμένη ο θεσμό και θέλω επίση να πω ότι η παρουσίαση του επενδυτικού πακέτου είναι καλό το ότι γίνεται εδώ. Εχθέ ελήφθησαν κάποιε αποφάσει και το σημερινό είναι ένα καλό δείγμα, ένα καλό μήνυμα ότι όλα αυτά γίνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο δικό μα το κόμμα, στο ΕΛΚ, κατά του τελευταίου μήνε είχαμε πολλά σημαντικά θέματα. Το πρώτο ήταν ότι είναι καλύτερα να ιδιωτικοποιηθεί το ιδιωτικό κεφάλαιο από το να αναλυφθούν νέα χρέη. Αυτή λοιπόν ήταν, ε, ήταν το οδηγό νήμα το οποίο μας οδήγησε τους τελευταίους μήνες. Better spending, καλύτερη εκπο... Ε, εκταμείευση κονδυλίων. Και η εμπειρία την οποία έχει ήδη συλλέξει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με την κινητοποίηση του ιδιωτικού κεφαλαίου, αυτή η εμπειρία είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Κύριε Χόια, γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στη μέθοδο που εφαρμόζουμε τώρα ε, έχει γύρει ένα-δύο θέματα. Παραδείγματο χάρη η αντικατάσταση. Δηλαδή προγράμματα που ήδη χρηματοδοτούνται θα συμπεριληφθούν σε αυτό το νέο πακέτο. Αυτό όμως δεν θα είναι σωστό. Επίσης γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε το ιδιωτικό κεφάλαιο σε νέα απόλυτα ασφαλή προγράμματα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε νέες επενδύσεις. Άρα υπάρχουν κάποια ερωτηματικά. Γνωρίζουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκκρεμούν κάποια θέματα ε, οι σημαντικέ αποφάσεις προφανώ και πρέπει να λαμβάνονται και από επιρρογνώμονε. όμως τα προγράμματα είναι πολιτικά. Πολιτικά πρέπει να συζητήσουμε. Και επιτρέψτε μου να πω προς το Συμβούλιο, για να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε αυτό το ιδιωτικό κεφάλαιο, Απευθύνομαι σε εσά, Συμβούλιο, επιτέλους να βοηθήσετε κι εσείς να σταματήσει αυτό το μπλοκάρισμα των ε, ε, διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό. Χρειαζόμαστε για την επόμενη χρονιά ένα σταθερό προϋπολογισμό για να μπορούμε να εφαρμόσουμε τα προγράμματά μας. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία, όπως σας είπα, οφείλουμε να ερευνήσουμε. Το δεύτερο που είναι σημαντικό για μας, ε, κυρίες και κύριοι, είναι το εξής. Το χρήμα μόνο του δεν μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα. Αυτό το είπε με απόλυτη σαφήνεια ήδη ο κύριος Γιούγκα. Κυρίε και κύριοι, οι επενδυτέ θα επανέλθουν στην Ευρώπη. Και σήμερα, αν δει κανεί επενδύσει, ε, το τι γίνεται στην Ευρώπη, βλέπουμε γίνονται επενδύσει στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία. Την προηγούμενη εβδομάδα πήγαμε στη Λετωνία. Συνάδελφοι, εκεί γίνονται επενδύσει. Μα γιατί γίνονται εκεί επενδύσει σήμερα, διότι αυτέ οι χώρε ε, τα τελευταία χρόνια προέβησαν σε μεταρρυθμιστικές αλλαγές μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της παγκοσμιοποίησης και να αλλάξουν ως κοινωνίες. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε περαιτέρω συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Οποτεδήποτε πρόκειται για τις τράπεζες, για τη ρύθμιση περίδιων κεφαλαίων, για την κοινή αγορά, ε, για τον ενεργειακό τομέα. Κοιτάξτε, στην ενέργεια δεν έχουμε κοινή αγορά, ούτε στον ψηφιακό τομέα. Μα γι' αυτό δεν γίνονται επενδύσεις. Αυτά λοιπόν είναι τα δικά μα τα καθήκοντα στην Ευρώπη, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Στην Ιταλία, α πούμε, που ουσιαστική ε, διαδρομή ε, ε, είναι ατέρμονη. Αυτό είναι πρόβλημα. Πώς να έχουν οι Ιταλοί επενδύσεις. Το ίδιο σχέδιο και για τη Γαλλία όταν άλλα προγράμματα προγραμματισμού όπως στη Γερμανία και αυτά είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα ε, δεν πρέπει κανείς να διρωτάται γιατί δεν γίνονται επενδύσεις άρα δηλαδή πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις το τρίτο θέμα που είναι σημαντικό για το ΕΛΚ για να υπάρχει κάποιο μέλλον στην Ήπειρό μας κυρίες και κύριοι θα το θίξω σήμερα ακροθυγός αλλά είναι πολύ σημαντικό πρόκειται για τη σταθερότητα των προπολογισμών που είναι ένα σύνεκουανόν για το να μπορέσουμε να επιτύχουμε ανάπτυξη εάν θέλουμε να, ε, να αποκομίσουμε τις σταθερότητα των αγορών. Εάν δεν επανήρχεται η κρίση, αυτό καταλαβαίνετε ότι ε, θα προκαλούσε περαιτέρω ζημιά στην Ευρώπη, άρα χρειαζόμαστε αξιοπιστία. Σήμερα ο κύριος Γιούγκερ μίλησε και παρουσίασε ένα πιστικό πρόγραμμα. Και παρακαλώ τους κίνσορες και τιμητές που θα εκφράσουν ήδη σήμερα την άποψή τους να έχουν κατά νου ότι οφείλουν να είναι επικοδομητικοί. Στην Ευρώπη έχουμε το πρόβλημα ότι όταν δεν υποβάλλει κανείς μία άποψη, αυτομάτως εμφανίζονται αυτούς που αποκάλεσα κίνσορες. Όμως, κυρίε και κύριοι, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι εκείνο που χρειαζόμαστε είναι να συμβάλλει κανείς, να πει «Ναι, καλή ιδέα, εγώ έχω μια ακόμα καλύτερη». Παρακαλώ λοιπόν να υπάρχει επικοδομητική κριτική, να υπάρχει αυτός ο πολιτισμός ε, της αισιοδοξία. Αυτό χρειαζόμαστε τώρα. Και αγαπητοί συνάδελφοι, απευθυνόμενο στο Συμβούλιο θέλω να πω το εξή. Τώρα ε, γίνονται οι προετοιμασίες για το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, Συμβούλιο Κορυφής. Και ανακύπτουν ερωτήματα όπως ε, δεν γίνονται πολλά, γίνονται πάρα πολύ λίγα. Σας παρακαλώ να συνειδητοποιήσετε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να στηρίξει τις υποχρώσεις της. Με τα 415 δις θα τηρήσουμε τις υποχρώσεις μας. Και εάν και οποτεδήποτε υπάρχουν προβλήματα σε κράτη-μέλη, είναι ανοιχτό το πρόγραμμα. Ελάτε να συζητήσουμε, ελάτε να δούμε το θέμα των επενδύσεων. Κυρίες και κύριοι, το ΕΛΚ στηρίζει το πρόγραμμα του κυρίου Γιούγκερ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς θέλουμε να εκπέμψουμε ένα μήνυμα νέα εκκίνησης. Σήμερα είναι μια πολύ καλή ημέρα για την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών το λόγο έχει ο πρόεδρος κύριος Πιτέλα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πριν από πέντε χρόνια αυτό το οποίο έλεγε η Επιτροπή Μπαρόζο ήταν σταθερότητα και λιτότητα. Εσείς όμως Πρόεδρε Γιούνκερ επιλέξατε να έρθετε εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σας ευχαριστούμε γι' αυτό για να παρουσιάσετε ένα σχέδιο επενδυτικό. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα πράγματα αλλάζουν. Απευθυνθήκατε προς επιχειρήσεις, προς τους πολίτες, προς τους σχολιαστές αν θέλετε τους πολιτικούς και αυτό το οποίο βλέπουμε πέρα από τις τεχνικές λεπτομέρειες είναι ότι το πνεύμα πλέον, το περιβάλλον αλλάζει. Πριν από πέντε χρόνια είχαμε αυτό τον τίτλο της λιτότητας. Αυτό που βλέπουμε φέτος είναι ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι επενδύσεις, η απασχόληση, η οικονομική ανάπτυξη. Πράγματι λάβατε κάποια μέτρα ήδη από την αρχή της νέας αυτής θητείας. Εμείς οι σοσιαλιστές λοιπόν θέλουμε να υποστηρίξουμε τη δέσμευσή σας αυτή και αυτό που θέλω να πω με περηφάνεια είναι το ακόλουθο, ότι η αλλαγή αυτή που ξεκινάει σήμερα είναι πραγματικά καρπός της πολιτικής μας μάχης. Πάρα πολλά στοιχεία μας πείθουν στα πλαίσια του σχεδίου αυτού, κυρίως η μέθοδος που θέλετε να ακολουθήσετε. Δεν μιλάμε πλέον για συμφωνίες οι οποίες γίνονται παρασκηνιακά ανάμεσα στις κυβερνήσεις. Για το νέο αυτό σχέδιο είδαμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμβάλλει άμεσα. Είπατε ότι δεν υπάρχει επιστροφή, δεν μπορούμε να πάμε πίσω. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να προωθήσουμε περισσότερε επενδύσει. Αυτό ζητούσαμε εδώ και πάρα πολλού μήνε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει προορατικό, προδραστικό ρόλο τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει ανάληψη κινδύνου στα πλαίσια των επενδύσεων αυτών. Χρειάζονται λοιπόν ακόμα και δημόσιοι πόροι προκειμένου να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν μα ενδιαφέρει τόσο πολύ η αξιολόγηση των οίκων αξιολόγηση. Αυτό που μα ενδιαφέρει περισσότερο είναι η ευημερία των ίδιων των πολιτών. Πόσο οι επενδύσει τελικά μπορούν να δημιουργήσουν θέσει απασχόληση. Και ήδη στο δικό μα ε, το πρόγραμμα, στη δική μα την ε, πρόταση οικονομική ανάπτυξη, την οποία απευθύναμε προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είπαμε ότι θέλουμε χρήσιμε επενδύσει. Κύριε Πρόεδρε, με απόλυτη ειλικρίνα λοιπόν θέλω να σας πω ότι πιστεύω ότι σήμερα ξεκινήσατε με μία σωστή μέθοδο. Αρχίζουμε και κινούμε στο σωστό δρόμο. Χρειαζόμαστε όμως ξεκάθαρες προτεραιότητες. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίσουν πού επενδύονται τα χρήματά τους και για τους πολίτες το πιο σημαντικό είναι η ενεργειακή μετάβαση, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες, πάρα πολλές χώρες που πλήττονται από τα φαινόμενα αυτά της κλιματικής αλλαγής. Σε καμία περίπτωση επίσης δεν μπορούμε να μεροληπτούμε. Πρέπει από κοινού να θέσουμε τη βάση για μια πραγματική βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτή είναι η αποστολή μας. Αυτή είναι η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πρέπει να προωθεί τα συμφέροντα των πολιτών. Θα πρέπει να λειτουργούμε ως κασάνδρες, αναφερόμενοι μόνο στις αρνητικές πτυχές του υφιστάμενου περιβάλλοντος το οποίο αντιμετωπίζουμε. Χρειαζόμαστε επίσης να καταφέρουμε να προωθήσουμε τις πρωταρχικές μας επενδύσεις, να καταφέρουμε να ξεμπλοκάρουμε, αν θέλετε, τις νέες αυτές επενδύσεις. Χρειαζόμαστε και τις τους απαραίτητους δημόσιους πόρους. Αυτά τα 20 δισεκατομμύρια στα οποία αναφερθήκαμε αρχικά αποτελούν μια πολύ καλή κοινή βάση. Θα πρέπει όμω να καταφέρουμε να θαρρύνουμε στη συνέχεια και τα κράτη-μέλη να συμβάλλουν και αυτά στο σχέδιο αυτό το οποίο παρουσιάσατε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο είπατε εντελώ ξεκάθαρα, κύριε Πρόεδρε, ότι οι συνεισφορέ των κρατών μελών δεν υπολογίζονται στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Δεν υπολογίζονται όσον αφορά το δημόσιο χρέο, δεν υπολογίζονται όσον αφορά το δημόσιο έλλειμμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακριβώ αυτή την ευελιξία χρειαζόμαστε στα πλαίσια του Συμφώνου. Γιατί ξέρω ότι στο παρελθόν δεν είχαμε καταφέρει να κάνουμε κάτι τέτοιο, επειδή υπήρχε αυτό το ταμπού των απόλυτων περιοριστικών όρων στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Θέλουμε να τηρήσουμε το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη, αλλά να το τηρήσουμε με τρόπο ευφύ, να έχουμε την απαραίτητη ευελιξία στα πλαίσια του προγράμματος αυτού. Εμείς είμαστε πολιτικοί ηθήνοντες, δεν λειτουργούμε ως λογιστές αυτή τη στιγμή. Κύριε Πρόεδρε, περιμένουμε λοιπόν τη δική σας ανακοίνωση όσον αφορά τη δυνατότητα ευελιξίας στα πλαίσια του συμφώνου αυτού. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα μέτρα και το έχουμε πει εμείς ξεκάθαρα ότι θέλουμε να έχουμε και τις απαραίτητες δημόσιες δαπάνες, δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες θα υποστηρίξουν τι εθνικέ οικονομίες και θα δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης χωρίς όμως να συνυπολογίζονται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ξέρω ότι θα πρέπει να αναλάβουμε κάποιο ρίσκο, κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ καλύτερο να κάνουμε κάτι τέτοιο από το να μετανοήσουμε εκ των υστέρων για πράγματα τα οποία δεν πράξαμε. Εμεί θα υποστηρίξουμε το σχεδιό σα, θα τον πλουτίσουμε τις δικές μας προτάσεις και θα σας ζητήσουμε ενδεχομένω στο μέλλον, όπως ήδη το είπατε, να το προωθήσουμε και να το επεκτείνουμε για άλλα τρία χρόνια. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην αρχή λοιπόν ενός νέου δρόμου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να εμφυσίσουμε δικαιοσύνη και ισοτιμία. Τα παιδιά στη Θεσσαλονίκη στα οποία αναφερθήκατε ή στα παιδιά της Μαδρίτης, στα οποία θα μπορούσα να αναφερθώ εγώ, είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρίσκονται σε ένα ισότιμο περιβάλλον ευημερία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τι ίδιε συνθήκε ακόμα και στη Λισαβόνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα δικά μα τα νοσοκομεία να βρίσκονται στην αιχμή του δόρατο όσον αφορά τι υποδοτέ, υποδομέ. Χρειαζόμαστε λοιπόν την απαραίτητο, το απαραίτητο όραμα, το απαραίτητο κουράγιο προκειμένου να κάνουμε αυτό το πράγμα πραγματικότητα. Σα ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρου ε, των, Ευρωπαίων Συντηρητικών Κοινωνιστών, ο κ. Καμάλ. Πρόεδρε, Juncker. Εμείς είμαστε μια ομάδα η οποία κοιτάει το μέλλον και όχι πίσω στο παρελθόν και ε, ε, πράγματι χρειάζεται να εξασφαλίσουμε ότι ε, θα έχουμε μια κάνουλα που θα ε, ποτίσει το μέλλον για να δημιουργηθεί ανάπτυξη και όχι να, χωρίς να πλημμυρίζει και να διώχνει τις επενδύσεις. Έχω μιλήσει με πολλούς ιδιωτικούς επενδυτές και τους έχω ρωτήσει τι τους εμποδίζει. Και την περασμένη εβδομάδα μίλουσα με ένα πολύ μεγάλο επένδυτη, πάνω από 600 εκατομμύρια λίρες επένδυη. Και μου λένε ότι τα κυβερνητικά προγράμματα είναι αστεία, δεν βλέπουν απόδοση σε αυτά. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν. Ε, μας ε, λένε ότι η κοινωτική νομοθεσία ε, παρεμποδίζει τις επενδύσεις. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Ένας παλιός ε, γερμανός ε, βιομηχάνος μου με ρωτούσε γιατί οι, μη, ε, οι, οι χώρες που είναι εκτός Ευρωζώνης είναι πιο ελκυστικές από τις χώρες της Ευρωζώνης για τις επενδύσεις. Μήπως το ευρώ λοιπόν είναι το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, το ερώτημα είναι πώς θα ξεμπλοκάρουμε μπλοκάρουμε αυτές τις επενδύσεις, ε, ε, πώς θα εξασφαλίσουμε, δεν μιλούμε μόνο για λεφτά, αλλά και για μεταρρυθμίσεις, όπως είπε ο κ. Βέμπερ. Να σας δώσω ένα-δύο παραδείγματα. Πριν μερικά χρόνια μιλούσαμε με μια βρετανική εταιρεία που ήθελε να επενδύσει στον Πρίντεζι της Ιταλίας. Χρειάστηκαν, ε, έχασαν 11 χρόνια για να δημιουργήσουν ένα τέρμιναλ υγροποιημένου φυσικού αερίου στον Πρίντεζι. 11 χρόνια έχασαν λόγω της γραφειοκρατίας. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι ε, αυτή η γραφειοκρατία δεν θα παρεμποδίσει τις επενδύσεις. Άλλο παράδειγμα. Εκατομμύρια ευρώ κρατικών κονδυλίων ε, στο, στο καινούργιο αεροδρόμιο της ε, Λιών και ακόμα δεν έχει ανοίξει. Ε, πώς λοιπόν θα ξεμπλοκάρουμε όλες αυτές τις επενδύσεις ε, χωρίς να βαρύνουμε τους ε, ε φορολογούμενους. Πώς θα αποφύγουμε τις καταστάσεις όπου ε, οι, ε, οι επενδύσεις θα οδηγούν σε απώλεια χρημάτων από τον των φορολογούμενων. Δώστε μας κάποιες λεπτομέρειες για αυτό το ταμείο, το ταμείο κύριε Γιούνκερ. Πέστε μας γιατί δεν επενδύουν αυτή τη στιγμή οι επενδυτές και τότε μπορεί να υποστηρίξουμε το σχέδιό σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρου των ε, ε, φιλελευθερών, ο κύριος Φεχόφστατ. Μα να σα πω επίση ότι δεν έχει ανοίξει καν το αεροδρόμιο του Βερολίνου. Άλλη ιστορία βέβαια αυτό. Εντάξει, ίσω το ίδιο πρόβλημα να έχουμε και εκεί. Είναι πάντως πάρα πολύ θετικό που έχουμε κύριε Γιούνκερ τη νέα σας αυτή πρόταση. Είπατε ότι θα ξεκινήσει να λειτουργεί την 1η Ιουνίου του 2015. Το νέο δηλαδή αυτό ταμείο μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί τότε. Αυτό είναι πολύ θετικό. Και για πέντε ολόκληρα χρόνια αγαπητοί συνάδελφοι Μιλάμε για εκατομμύρια, μιλάμε για project bonds. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα συγκεκριμένο ποσό μπροστά μας και μιλάμε πραγματικά για το επενδυτικό αυτό χάσμα, το οποίο είναι τεράστιο, 700 δισεκατομμύρια ευρώ. Από την αρχή της κρίσης μειώθηκαν οι επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 14% ε, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες καθόλου αυτό το πενταετές διάστημα οι επενδύσεις παρέμειναν σταθερές. Το ζήτημα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τρει παρατηρήσεις λοιπόν θέλουμε να κάνουμε, προκειμένου το σχέδιο αυτό να λειτουργήσει ομαλά. Πρώτον, αυτό το επενδυτικό σχέδιο, κύριε Γιούνκερ, δεν μπορεί να εξεταστεί ξεχωριστά από άλλες πολιτικές. Ήδη από τις αρχές του 2015, όταν προτείνεται νέα νομοθεσία, η νέα αυτή νομοθεσία δεν θα πρέπει να αφορά μόνο το ζήτημα αυτό, αλλά αν θέλετε και τι συμπληρωματικέ εκείνε πολιτικέ που είναι απαραίτητε. Πρώτον, πρέπει να γίνουν προφανώ οι διαφορετικέ μεταρρυθμίσει στα κράτη-μέλη. Ο κύριο Βέμπερ έδωσε κάποια παραδείγματα, αγορά εργασία, συντάξει και το καθεξής. Και δεν μπορούμε να μιλάμε καν για ρεσιμότητα αυτή τη στιγμή, οι προϋποθέσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε επενδύσεις αν δεν υπάρχει το απαραίτητο ασφαλές περιβάλλον. Πρέπει τα κράτη-μέλη να κάνουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις προκειμένου να προσελκύσουν επενδύσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να ενταχθεί και η διάσταση της αιρεσιμότητας, των προϋποθέσεων δηλαδή για να γίνουν οι επενδύσεις αυτές ήδη από την αρχή του 2015. Επίσης, δεύτερη πτυχή του προγράμματο αυτού θα πρέπει να είναι το ότι θα πρέπει το πρόγραμμα να είναι ανοιχτό προ διάφορε αγορέ, την ενεργειακή αγορά, την ψηφιακή αγορά και το καθεξής. Δεν αρκεί απλώς να έχουμε μια διασύνδεση ανάμεσα στην Ισπανία και τη Γαλλία όσον αφορά την ενέργεια, αν στη Γαλλία υπάρχει μια νομοθεσία η οποία θα μπλοκάρει μια τέτοια επένδυση, αν στη Γαλλία υπάρχει μια νομοθεσία που δεν επιτρέπει την εισαγωγή ενέργειας από την Ισπανία. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και στην ψηφιακή αγορά. Αν συνεχίσουμε να έχουμε 28 διαφορετικού επιθεωρητέ όσον αφορά την ψηφιακή αγορά, ξεχάστε αυτό το περιβόητο ευρυζωνικό κοινό περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι δεν θα υπάρχουν όλοι αυτοί οι περιορισμοί, ότι δεν θα υπάρχει ο κατακαιρματισμό. Όσον αφορά τι ε, κεφαλαγορέ, και βλέπω τον κύριο Χίλ, τον επίτροπο εδώ μαζί μα, αν θέλουμε πραγματικά ενοποίηση των κεφαλαγορών, κύριε επίτροπε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί και εκεί να υπάρχει διασύνδεση ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Να μπορούμε να έχουμε πιστώσει μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιταλία, για παράδειγμα. Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν απλώ και μόνο ένα επενδυτικό σχέδιο. Χρειαζόμαστε και ένα γενικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο που θενοποιήσει όλε αυτέ τι διαφορετικέ τομεακέ αγορέ που εξαρτώνται από το επενδυτικό σα σχέδιο, κύριε Γιούγκερ. Τέλο, όσον αφορά τη λειτουργία του Ταμείου αυτού καθεαυτό. Α είμαστε ειλικρινεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο εμπλοκής δημοσίων χρημάτων. Έχουμε μόνο δημόσιο χρέος. Δημόσια χρήματα διαθέσιμα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιηθεί ένα σύστημα εγγύσεων, ένα σχέδιο εγγύσεων. Για τις εγγύσει δεν χρειάζεστε κεφάλαιο, μπορείτε να δημιουργήσετε χρήματα μέσω μόχλευσης και το πιο σημαντικό κύριε Πρόεδρε, είναι να ασχοληθεί όμω και η άλλη πλευρά, όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προφανώ θέλει να προωθήσει το πρόγραμμα αυτό, δικό σα είναι άλλωστε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εμπλακεί και το Συμβούλιο και τα 28 κράτη-μέλη. Αν τα 28 κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση εμπλακούν στο δικό σα το σχέδιο και συνεργαστούν, κύριε Πρόεδρε, τότε πραγματικά θα έχετε ένα πολύ καλύτερο σύστημα εγγύσεων από τα χρήματα αυτά τα οποία έχουμε διαθέσιμα αυτή τη στιγμή. Και να ζητήσω από τον κύριο Γκότσι να θέσει το ζήτημα αυτό στο επόμενο Συμβούλιο, στο οποίο θα προεδρεύσει η Ιταλική κυβέρνηση τον Δεκέμβριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεισφέρει σε αυτό το σύστημα εγγυήσεων κάθε κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να προωθήσουμε τι επενδύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο πρέπει να προωθήσει, κύριε Γκότση, η Ιταλική Προεδρία. Και για ποιο λόγο να μην προβλέψουμε και φορολογικέ απαλλαγέ κύριε Πρόεδρε. Θα μπορούσε κάθε κράτος μέλος προωθώντας ένα τέτοιο μέτρο να καταφέρει να συμβάλλει ακόμα περισσότερο. Θα μπορούσαν για παράδειγμα τα κράτη-μέλη να μην επιβάλλουν και σύστημα φορολογίας το οποίο θα συνοδεύει το ταμείο αυτό και τη χρηματοδότηση από αυτό το ταμείο. Κατά αυτόν τον τρόπο θα κινητοποιηθούν και πολλοί άλλοι επενδυτές, όχι μόνο θεσμικοί επενδυτές αλλά και επενδυτές από τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρετε ότι αν, υπάρχουν, ε, αν υπάρχει μια πάρα πολύ αυστηρή φορολογία, υπάρχουν πάρα πολλοί οποίοι θα αποθαρρυνθούν. Αντίθετα, αν προβλέψουμε το απαραίτητο καθεστώς φοροαπαλλαγών, τότε θα κινητοποιήσουμε πάρα πολλού νέου επενδυτέ Και ολοκληρώνοντα, κύριε Πρόεδρε, Ας μην προσπαθήσουμε αυτή τη στιγμή να ικανοποιήσουμε ξεχωριστά τις επιθυμίες και τις προσδοκίες κάθε κράτους μέλου ξεχωριστά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αντίθετα να προωθήσουμε τη βούληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και πιστεύω ότι από κοινού θα καταφέρουν να προωθήσουν σημαντικότερε επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Εκ ο Παρακαλώ το περίφημο πακέτο των 300 δισεκατομμυρίων ευρώ που μας υποσχεθήκατε στις 15 Ιουλίου είναι άδειο. Είναι σταγόνα στον ωκεανό. Τι μας παρουσιάσατε 15 δις από τον κοινοτικό προϋπολογισμό 16 δις και 5 δις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ούτε ένα ευρώ φρέσκο χρήμα. Και μας υπόσχεστε ότι θα πετύχετε μόχλευση 15 φορές, 1 προς 15. Δεν υπάρχει ένας οικονομολόγος στον κόσμο που να πιστεύει ότι σε συνθήκες στασιμότητας της οικονομίας με τον κίνδυνο μιας νέας ύφεσης στην ευρωζώνη και με τον κίνδυνο του αποπληθωρισμού είναι δυνατόν κεφάλαια να μοχλευτούν 15 φορές. Ακόμη και οι Υπουργοί Οικονομικών που σας υποστηρίζουν και μετέχουν στις ομάδες που λένε ζήτω το πακέτο juncker σας λένε χρειάζεται φρέσκο χρήμα χρειάζονται νέα κεφάλαια και η ιστορία της παγκόσμιας οικονομίας λέει ότι σε εποχές στασιμότητας ή και ύφεσης χωρίς ισχυρούς δημόσιους πόρους δεν είναι δυνατόν να υπάρξει στροφή στην ανάπτυξη. είπε ο κύριος Φέρχοφστατ ότι οι επενδύσεις στην ευρωζώνη μετά την κρίση είναι 15 φορές παρακάτω ενώ στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι παραπάνω. Γιατί, γιατί εκεί έριξαν χρήμα, γιατί εκεί η, τράπεζα έπαιξε ένα αναπτυξιακό ρόλο. Εσείς εδώ δεν αλλάζετε τα εργαλεία. Κύριε Γιούγκερ, κάποια στιγμή προτείνατε να αξιοποιηθεί και ένα μέρος από τα λιμνάζοντα 500 δισεκατομμύρια ευρώ του ESM μόλις ο κύριος Σόιμπλε είπε όχι και έβαλε το γερμανικό βέτο, το ξεχάσατε. Θα μας πείτε κάτι για αυτή την πρόταση. Και επειδή αναφερθήκατε και στα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη, από την πατρίδα μου, η δική σας πολιτική με την Τρόικα έχει προκαλέσει ύφεση 25%, ανεργία 30%, ανεργία στους νέους 60%, ανθρωπιστική κρίση το περίφημο πακέτο σας είναι business as usual σε μια λογική γερμανοκρατούμενης ευρώπης και σκληρής μονόπλευρης λιτότητας. Εκ μέρους των Πρασίνων, ο πρόεδρος κύριος Λάμπερτς. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιούνκερ που ήρθατε τόσο γρήγορα, ε, ένα μήνα μετά εδώ, για να μας παρουσιάσετε αυτό που αρχίζει να φαίνεται ως να μοιάζει με ε, πρόγραμμα επενδύσεων. Ε, τηρήσατε λοιπόν την υπόσχεσή σας. Συμφωνούμε με την διάγνωσή σας ότι λείπουν οι επενδύσει. Όμως τι εννοούμε με τη λέξη επενδύσεις. Για μα επενδύσεις δεν είναι αυτά τα κονδύλια τα οποία οποία για βραχυχρόνια παίζονται κάπου και στοιχηματίζονται. Δεν είναι αυτοί οι επενδυτές. Ε, επενδύσεις δεν είναι, επίσης δεν καλύπτουν ε, ως ο όρος τις διάφορες φούσκες ε, που βλέπουμε στην Ευρώπη τη μία μετά την άλλη. Να διαδέχονται τη μία μετά την άλλη. Επενδύσεις ε, δεν σημαίνουν επίσης ε, δισεκατομμύρια για να δημιουργηθεί ένα ε, ένας πυρηνικός σταθμός εδώ, ένα αεροδρόμιο εκεί που δεν θα υπηρετεί κανένα ή να γεμίσουμε με μπετόν την πρωτεύουσα της Ιρλανδίας ή τις παραλίες της Ισπανίας. Δεν μιλάμε για τέτοιου είδου επενδύσει, ούτε για επενδύσει που έχουν στο μυαλό του μόνο το κέρδο. Η μόνη χρήσιμη επένδυση είναι η ανθρώπινη, υλική οικονομική ε, επένδυση ε, που θα εξασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια που γίνεται με αυτό το στόχο. Μιλούμε για την οικολογική μεταρρύθμιση, ε, μιλούμε για την κοινωνική συνοχή, μιλούμε για την κατάρτιση και την εκπαίδευση, για την έρευνα. Αυτή πρέπει να είναι η προορισμοί των επενδύσεων. Και το σχέδιό σας ε, περιλαμβάνει ένα αριθμό αυτούς τους στόχους. Όμως από πλευράς όγκου και συνολικού κεφαλαίου, τα 21 δισεκατομμύρια τα οποία δεν είναι φρέσκο χρήμα, δεν πιστεύουμε ότι θα είναι επαρκή για να δημιουργήσουν μόχλευση 350 δις. 315 δις. Και μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για χρήματα τα οποία ήδη υπάρχουν. Τα αφαιρούμε από άλλα προγράμματα, όπως για παράδειγμα προγράμματα έρευνας. Δεν νομίζω ότι είναι, αυτό, είναι ότι είναι σωστό αυτό. Είναι σαν να πριονίζουμε το κλάδι που καθόμαστε. Το σχέδιο αυτό θέλει να ε, επιτρέψει στο δημόσιο, στον κρατικό τομέα να καλύψει τις πρώτες ε, ζημίε μια επένδυση. Τι σημαίνει όμω αυτό, Είναι δυνατόν να καλύπτουμε εμεί τι ζημίε ε, του ιδιωτικού τομέα και μετά τα κέρδη να επιστρέφουν στο ιδιωτικό τομέα, Είναι σωστό αυτό. Τώρα, αν μπορέσουμε να βελτιώσουμε το σχέδιο, θα συνεισφέρουμε επικοδομητικά. Αλλά να υπογραμμίσω κάποια μέτρα τα οποία λείπουν και θα μπορούσαν να το συμπληρώσουν. Πρώτον, να κλείσουν τα καζίνο. Οι επενδυτικές αποφάσεις λαμβάνονται μέσω σύγκριση. Όσο έχουμε τη δυνατότητα οι επενδυτές να δημιουργούν καζίνο και, να, ε, και μάλιστα με κρατικές ε, επενδύσεις και να κερδίζουν έτσι χρήματα, θα κάνουν αυτό. Θα πρέπει να τα κλείσουμε λοιπόν. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ ε, δόθηκαν για πυρηνικούς σταθμούς και ελάχιστα για την πραγματική οικονομία. Μετά, καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής. 21 δισεκατομμύρια ευρώ θα είχαν ήδη ε, πληρώσει κάποιες πολυεθνικές αν πλήρωναν φόρους όπως θα έπρεπε να πληρώνουν. Συνεπώς, θα πρέπει η φοροδιαφυγή, η καταπολέμηση φοροδιαφυγής της, φορο... της φορολογικής απάτης να συμπεριληφθεί. Επίσης, ε, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να ε, μειώσουμε, να ε, επανακατευθύνουμε τις ε, επιδοτήσεις που δίνουμε στην, στο πετρέλαιο και στην πετρελαϊκό τομέα. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ αυτή τη στιγμή χρηματοδοτούμε ημερησίω με ένα δισεκατομμύριο ευρώ τον Πούτιν και τι αραβικέ χώρες. Ευχαριστώ. Die e Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι ε, χρησιμοποιούσαμε σημαντικότατη μόχλευση στο City του Λονδίνου, αλλά οχριά η μόχλευση αυτή απέναντι στη μόχλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς δεν έχουμε αυτά τα 350 δισεκατομμύρια ευρώ και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν κάνετε σωστές επιλογές. Όπως είπε ο Ασά, η Ευρωζώνη βρίσκεται σε συνεχή κατάσταση και έχει συνεχή στάση στασιμότητας. Προσπαθείτε εσείς να εφαρμόσετε κύριε Γιούνκερ αυτή τη στιγμή μία θαραλέα λύση, αλλά παρόλα αυτά η βάση δεν είναι η σωστή αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι θα καταφέρουμε αυτή τη στιγμή με το πρόγραμμά σας αυτό να οδηγηθούμε στην ανάπτυξη την οποία προτείνατε. Δεν θα καταφέρουμε να προστατεύσουμε την οικονομική δραστηριότητα σε πλαίσιο αντικσοτήτων. Νομίζω ότι μετά την κρίση του 2008 είχαμε πάρα πολλέ απώλειε στον Ηνωμένο Βασίλειο και αντίστοιχα έχουμε δει στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση πάρα πολλέ χώρε όπω η Ισπανία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία οι οποίε επλήγησαν από την οικονομική κρίση. Βέβαια η Γερμανία έχει πολύ καλέ βιομηχανικέ σχέσει, τι πάρα πολύ καλέ θετικέ υποδομές οι οποίε χρειαζόμαστε την απαραίτητη οικονομία κλίμακο, καθώ επίση και τι σημαντικότατε εταιρείε στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί λοιπόν να κινηθεί πάρα πολύ θετικά. Θεωρώ όμω ότι δεν μπορούν να ισχύουν ανάλογε συνθήκε σε όλε τι υπόλοιπε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Νότια ιδίω Ευρώπη είναι πραγματικά όνειδο το ότι έχουμε ένα τέτοιο υψηλότατο ποσοστό ανεργία. Δεν μπορείτε να λέτε αυτή τη στιγμή ότι μπορούν να κινηθούν με τον ίδιο ρυθμό και με τον ίδιο τρόπο οι χώρε τη Νότια Ευρώπη. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι εξαιτία του ευρώ υπάρχουν αποπληθωριστικέ τάσει παντού στη Νότιο Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι ούτε τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ, ούτε η μόχλευση η οποία προτείνεται και θα οδηγεί στα 315 δισεκατομμύρια ευρώ θα επιφέρει κάποια ουσιαστική λύση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να προστατεύσουμε του πολίτε, να εγγυηθούμε το μέλλον τους. Δεν νομίζω ότι έχουν έρθει νωρίτερα τα Χριστούγεννα, κύριε, ε, κύριε Γιούνκερ. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που μας προτείνεται είναι μία άλλη σφαλμένη λύση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Το λόγο λοιπόν έχει τώρα ο κύριος Άνεμανς εκ μέρους ε, των ε, ε, μη εγγεγραμμένων. Κύριε Γιούνκερ, δεν νομίζω ότι υπερβάλλω ισχυριζόμενος ότι το πακέτο της ανάπτυξης και της απασχόλησης είναι μία φάρσα. Είναι απλά ε, μία σειραφή διαφόρων πραγμάτων τάκτος ερημένων και απλά ε, σε αυτό το συμπίλημα έχει τοποθετηθεί μία ετικέτα. Όλα αυτά λοιπόν είναι άχρηστα και ούμονον αυτό, αλλά όλα αυτά κάτω από το μανδύα της μόχλευσης. Υποτίθεται ε, τα ποσά, το ποσό, τα 315 δισεκατομμύρια ε, θα επιμεριστούν στα κράτη-μέλη Αμπεμπαμπλόμ, αυτό το παιχνιδάκι νομίζω θα μπορούσαμε να παίξουμε ως παιδιά, αλλά ξέρετε κύριε Γιούνκερ ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ότι δυστυχώς ε, και εσείς έχετε τα προβλήματά σας, ε, έχετε τα σκάνδαλα που σας ε, απασχολούν, η Κομισιόν έχει ήδη αμαυρωθεί και κατόπιν τούτου οφείλουμε να πούμε το εξής αντιμετωπίζετε πράγματι ένα τεράστιο πρόβλημα. Το πρόβλημά σας είναι ότι χάσατε την αξιοπιστία σας και τελικά έχουμε ένα πρόεδρο ε, τον οποίο δεν μπορούμε καθόλου να εμπιστευτούμε. Εκ μέρους λοιπόν ε, του Συμβουλίου, ο Υπουργός κύριος Παντουάν. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, αγαπητέ Πρόεδρε της Επιτροπής. Η πρωτοβουλία του Προέδρου κ. Γιούγκερ είναι μη τι άλλο επίκαιρη. Ε, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η ανάπτυξη στην Ευρώπη δεν είναι ικανοποιητική. Υπάρχουν ε, προβλέψεις ε, σχετικά με την ανάπτυξη που έχουν μια καθοδική τάση. Υπάρχει λοιπόν σοβαρός κίνδυνος να μετακινηθούμε προς την στασιμότητα ενώ η ο πληθωρισμός παραμένει πολύ χαμηλός. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να υπάρξει ανάπτυξη. Απομακρύνεται, θα έπρεπε να απομακρύνουμε την στασιμότητα. Αυτό είναι απαραίτητο για ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ιταλική Προεδρία στο Συμβούλιο έχει θέσει την στροφή προς την απασχόληση στο επίκεντρο των προσπαθειών της. Και είπαμε ότι είναι τρεις οι απαραίτητοι πυλώνες. Να υπάρξει αλλαγή των υποδομών, η Ευρώπη να στραφεί προς τα έξω και να στηριχθούν οι επενδύσεις. Η ανάπτυξη των επενδύσεων είναι καθοριστική καθοριστική σημασία έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπει σε ένα νέο δρόμο ανάπτυξη. Οι επενδύσει μάλιστα στηρίζουν ε, τη ζήτηση ε, και επίση μπορούν να δώσουν και τη δυνατότητα να υπάρξει κάποια ισορροπία ανάμεσα σε ζήτηση και ε, προσφορά. Όπω είπαν και πάρα πολλοί, τα τελευταία χρόνια η πτώση των επενδύσεων ήταν τραγική, γενικευμένη. Τώρα πλέον πρέπει να αντιστρέψουμε αυτή την τάση. Οι μεταρρυθμίσει στι υποδομέ είναι απαραίτητε σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι μεταρρυθμίσει θα βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, θα υπάρχουν καλύτερες προοπτικές για επενδύσεις και κέρδος. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα σε κάποια κράτη-μέλη είχαν αυτομάτως ένα spill-over effect, όπως λέγεται, μετακυλήθηκαν θετικές επιπτώσεις σε άλλα κράτη-μέλη. Αρκεί να έχουμε κατά νου και την Τραπεζική Ένωση, όπως επίσης ε, και αυτά που αποφασίστηκαν πρόσφατα για την αυτόμαντη ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικό επίπεδο. Όλα αυτά αλλάζουν τους κανόνες, αλλάζουν τις συμπεριφορές και τους πόρες. Η ε, ολοκλήρωση δίνει δυνατότητα για τις επενδύσεις ε, και αυτό μπορεί να γίνει, μπορεί να είναι εφικτό. Το δίλημα το οποίο αντιμετωπίζει κανείς συχνά, κατά πόσον είναι απαραίτητο να υπάρχει περισσότερο χρήμα ή περισσότερα προγράμματα, είναι λάθος δίλημα. Ισχύουν και τα δύο. Αν υπάρχουν προγράμματα που είναι καλά, μπορούν να αυξηθούν και οι πόροι άμεσα ή έμεσα αυτό που είναι απαραίτητο για την οικονομία. Η επιτελική ομάδα για τις επενδύσεις ε, που θέσπισε ε, το ΕΚΟΦΗΝ και εκεί συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κρατημέλη. Αυτή η ομάδα έχει ήδη δώσει συγκεκριμένα αποτελάσματα για οικονομικά προγράμματα. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση για το μέλλον. Το πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε ο πρόεδρος Επιτροπής μπορεί να δερματίσει καθοριστικό ρόλο έτσι ώστε να δοθεί όθηση στις επενδύσεις, στην ανάπτυξη, να δρομολογηθεί μια διαδικασία που μπορεί να ενισχυθεί εν ευθέτω χρόνο μια διαδικασία που θα συνδέεται περισσότερο και με άλλες πολιτικές ε, που διαθέτει η Ευρώπη ή που θέλει να υιοθετήσει. Το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ προτίθεται να δώσει μια θετική όθηση ε, ήδη τις αμέσως επόμενες ημέρες. Είναι επίση απαραίτητο και νομίζω αυτό το είπανε πάρα πολύ να ε, δραστηριοποιηθούν τόσο ιδιωτικές επενδύσεις όσο και οι δημόσιες. Είναι σημαντικό οι δημόσιοι πόροι να κινητοποιηθούν έτσι ώστε να υπάρχει η μόχλευση των ιδιωτικών κεφαλαίων να ε, δοθεί δυνατότητα ανάληψης κινδύνων. Αλλά μην ξεχνάμε ότι οι δημόσιες επενδύσεις έχουν και άμεσες επιπτώσεις θετικές στις ιδιωτικές επενδύσεις, κυρίως ε, όσον αφορά ε, τις περιόδους όπου υπάρχει χαμηλή ζήτηση. Το θέμα της ασθενούς σφαιρικής συνολικής ζήτησης, όπως ισχύει τώρα, είναι κάτι που επηρεάζει επιχειρήσεις, αποδυναμώνει την εμπιστοσύνη, άρα δηλαδή αυξάνονται οι κίνδυνοι των επενδύσεων. Βρισκόμαστε μπροστά σε κίνδυνο κατάρρευσης αγορά, γι' αυτό λοιπόν ο δημόσιο ταμέας θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί από κοινού με τον ιδιωτικό. Και για να υπάρχουν ιδιωτικέ επενδύσει, το επαναλαμβάνω, είναι απαραίτητο να υπάρξουν μεταρρυθμίσει, πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον και επίση να εισαχθούν και νέα χρηματοπιστωτικά εργαλεία. Αυτή την προοπτική τη βλέπω να συνδέεται με μια ιδέα που προκύπτει από την περίφημη Ένωση, Κεφαλουχική Ένωση, μαζί με την Τραπεζική Ένωση και την κινητοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων. Θα πρέπει να βρούμε και άλλα εργαλεία τα οποία ενισχύουν αυτά που ήδη υπάρχουν. Σε όλα αυτά λοιπόν είναι είναι σημαντικός ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και σε συνεργασία με τις Εθνικές Τράπεζες Ανάπτυξης θα πρέπει η συνεργασία να ενισχυθεί. Είναι ισχυρή αλλά να ενισχυθεί περαιτέρω έτσι ώστε όλοι μαζί να προσπαθήσουν όχι μόνο να πολλαπλασιαστούν οι πόροι αλλά να πολλαπλασιαστεί και η τεχνική δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων και ως εκ τούτου κατεύθυνση ε, των κονδυλίων σε σωστά προγράμματα. Στρατηγικά ε, γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει ανάπτυξη και στον ενεργειακό τομέα και σε πολλούς άλλους σημαντικούς. Σημαντική αυτή η τομή, αλλά είναι σημαντική στο σύνολό τους δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η σταδιακή μείωση των επενδύσεων στην Ευρώπη είναι εκείνη που οδηγεί στο να απομακρύνεται η Ευρώπη από το τεχνολογικό υψηλό επίπεδο. Και έτσι δεν προκύπτει και ανάπτυξη. Ε, τελειώνοντας, ε, θέλω να εκφράσω το εξής. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν ταχύτατα. Οι προοπτικές ε, των Ευρωπαίων, στην, των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλύτερες, αλλά ελοχεύει ακόμα και αυξάνεται και ο κίνδυνος της απογοήτευσης. Σήμερα το πρόγραμμα που παρουσίασε η Επιτροπή είναι σημαντικό, απαιτεί βέβαια κάποιο χρόνο περαιτέρω για να ολοκληρωθεί, να ελεγχθεί. Εν τω μεταξύ μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα επιλεγμένα προγράμματα, μπορούμε να κατευθύνουμε τους υπάρχοντες πόρους προς αυτά τα προγράμματα, μπορούμε από κοινού να δώσουμε ένα μήνυμα εμπιστοσύνη ε, εμπιστοσύνη λοιπόν από πλευρά του κοινού τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αντιστρέψουμε την φθήνουσα τάση των ιδιωτικών επενδύσεων. Οι ε, προοπτικές ανάπτυξης που είναι χαμηλές ε, σε μεγάλο βαθμό εξηγούν και το ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη προς τους πολιτικούς εκ μέρους των Ευρωπαίων πολιτών. Και αυτό είναι καθήκον των θεσμών. Είμαι λοιπόν πεπισμένος ότι η πρωτοβουλία που παρουσιάστηκε σήμερα εκ του κυρίου κυρίου Γιούνκερ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι παρά μόνο το πρώτο βήμα σημαντικό σε αυτή την οικονομική αλλαγή που πρέπει να επέλθει και ως εκ τούτου και στη δυνατότητα της Ευρώπης να προσφέρει και πάλι ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πάντοβαν και τελειώνοντας θα ήθελα να δώσω το λόγο εκ μέρους Επιτροπής στον Αντιπρόεδρο κύριο Κατάινεν. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω ήδη όλους για τις ε, πολύτιμες απόψεις που εκφράσατε. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να συγκεντρωθούμε στην ε, στενή συνεργασία έτσι ώστε το σχέδιο αυτό να υλοποιηθεί. Σήμερα η Επιτροπή Juncker ικανοποιεί την πρώτη υπόσχεση που έδωσε όταν διορίστηκε. Υποβάλλει ένα πρόγραμμα επενδύσεων που θα αλλάξει τον τρόπο χρήση των κρατικών κονδυλίων για επενδύσει στην Ευρώπη. Υπάρχει ρευστότητα στην αγορά. Τα ε, επιτόκια είναι πολύ χαμηλά και οι αγορέ έχουν σταθεροποιηθεί. Ταυτόχρονα υπάρχει και σημαντική ε, ανάγκη και ζήτηση για αξιόπιστα επενδυτικά σχέδια. Παρ' όλα αυτά δεν γίνονται επενδύσει. Υπάρχει δηλαδή ένα μεγάλο χάσμα ανάμεσα στην πραγματικότητα και στη θεωρία οι κρατικέ αρχές μπορούν να παίξουν ένα πιο δραστήριο ρόλο και στην πλευρά τη ζήτηση και στην πλευρά τη προσφοράς. Χρειαζόμαστε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για project. Project τα οποία θα ε, υπηρετούν τις, ε, τους μακροπρόθεσμους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταφορές, ενέργεια, περιβάλλον ε, κλπ. Η Ευρώπη πρέπει να είναι ενωμένη και καινοτόμα. Μόνο έτσι θα μπορέσει να υλοποιηθεί ένα τέτοιο project. Χρειάζεται ισχυρή πολιτική στήριξη και βασιζόμαστε στη στήριξή σας έτσι ώστε να διατηρήσουμε τη φιλοδοξία αυτού του, του, αυτής της πρότασης και να στείλουμε το μήνυμα ότι η φωνή σας ακούστηκε. Ε, σε ό,τι αφορά την ε, πρόσθετη ε, κινητοποίηση κεφαλαίων. Ε, είναι σημαντικό αυτό το θέμα, αλλά δεν είναι επαρκής η απλή συζήτησή του. Δεν είναι το θέμα να βάλουμε απλώς νούμερα στο τραπέζι. Εμείς υποβάλουμε ένα πρόγραμμα σημαντικής μεταρρύθμισης, ριζικής μεταρρύθμισης και θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι πραγματικέ επενδύσει θα γίνονται στην πραγματική οικονομία και ότι θα δημιουργήσουν καινούριε θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη. Το ε, επενδυτικό πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα τρίγωνο με τρία κομμάτια, τρει πλευρέ. Πρώτον, θα εξασφαλίσουμε ότι οποιοδήποτε ευρώ επενδύεται μέσω αυτού του προγράμματο θα έχει τη μέγιστη δυνατή, ε, ε, ε, το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στην οικονομία. Αυτό θα το πετύχουμε συνεργαζόμενοι με την ΕΤΕΠ. Το ταμείο αυτό θα χρηματοδοτηθεί και από την ΕΤΕΠ και από τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση με 21 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα νέα φρέσκα κεφάλαια θα είναι πάνω από 60 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία θα πάνε στην πραγματική οικονομία. Με αυτά θα χρηματοδοτήσουμε και θα δανείσουμε. Θα χρηματοδοτήσουμε project ε, σύγχρονα. Και τα χρήματα αυτά θα δώσουν εγγυήσεις σε project υψηλού κινδύνου ε, έτσι ώστε να συμπληρώσουμε τις, ε, τη χρηματοδότηση που θα από την ΕΤΕΠ. Επίσης, θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση μακρο, μακρόπνοων επενδυτικών στρατηγικών και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το Ταμείο θα φέρει καινούργια χρήματα και από ιδιωτικούς επενδυτές, οι οποίοι θα έχουν να αντιμετωπίσουν μικρότερο κίνδυνο. Αυτό το πολλαπλασιαστικό φαινόμενο θα ε, επιτρέψει να ρεύσουν πάνω από 300 δισεκατομμύρια ευρώ στην πραγματική οικονομία. Πρόκειται μάλιστα για ένα συντηρητικό σενάριο που βασίζεται σε παλιότερες εμπειρίες μας και τις εμπειρίες της ΕΤΕΠ. Δεν μιλάμε για σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Ε, κάποιοι λένε ότι δεν πρόκειται για πραγματικό χρήμα. Α, όλα αυτά είναι ανοησίες κατά την άποψή μου. Πρόκειται για πραγματική πρόσθετη δυνατότητα χρηματοδότησης πάνω από 60 δισεκατομμύρια ευρώ με, με ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτά, αυτά τα χρήματα θα δημιουργήσουν καινούριε θέσει εργασία και καινούριε επένδυσεις. Δεν μοιράζουμε χρήματα με τρόπο που να πλήττουν τους προπολογισμού μας και τα, τα, δημόσια οικονομικά. Εμείς κάναμε το καθήκον μας. Το επόμενο βήμα είναι κυβερνήσεις να στηρίξουν το σχέδιο και να συνεισφέρουν και αυτές με ποσά από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Οι συνεισφορές των εθνικών κρατών μελών θα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Επίσης, περιμένουμε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν καλύτερα τα ευρωπαϊκά διαφορετικά ταμεία και να διπλασιάσουν την ε, χρήση εγγυήσεων και δανείων. Αυτή τη στιγμή το 92% των διαφορετικών ταμείων ε, ε, ε, χρησιμοποιούνται και μετά τα ξεχνάμε. Θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε καλύτερα αυτά τα ποσά. Με τρόπο ώστε να επηρεάσουμε την πραγματική οικονομία. Στο κέντρο, στην καρδιά αυτού του πακέτου όμως υπάρχει μια πολιτική επιλογή. Ή θα συνεχίσουμε την πεπατημένη με τα παραδοσιακά δάνεια κλπ. Ή θα χρησιμοποιήσουμε τον προπολογισμό μα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, έτσι ώστε να υποστηρίξουμε αυτού που παίρνουν ρίσκο και να αυξήσουμε τη δανειοδοτική ικανότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι μάλιστα η επιλογή που κάναμε εμεί. Είναι μια καινούρια προσέγγιση. Να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δημόσια κονδύλια, τα κρατικά κονδύλια. Θέλουμε αυτά τα χρήματα να φτάσουν στην πραγματική οικονομία. Μαζί με την ΕΤΕΠ δημιουργούμε ε, μια ε, ένα, το, μάλλον ε, με διαφάνεια τον ε, θεσμό του έμπιστου αξιόπιστου επενδυτή. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και τα εργαλεία των κρατών μελών καλύτερα. Αυτό ζητούν οι επενδυτέ. Υπάρχει ρευστότητα εκεί έξω. Αλλά οι επενδυτέ μα λένε χρειάζονται καλά διατυπωμένα, ψηλή ποιότητα project. Η Task Force της Κομισιόν για τη ΣΕΤΕΠ μαζί με τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή εντοπίζει πάνω από χίλια project τα οποία θα αξιολογηθούν. Θέλουμε να ε, βάλουμε μια ευρωπαϊκή σφραγίδα για τα πιο αξιόπιστα από αυτά. Χρειαζόμαστε επενδύσεις για το μέλλον. Ε, δεν χρειαζόμαστε άλλες φούσκες. Γι' αυτό το λόγο προτείνουμε το συνδυασμό εγγύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο με, ε, μαζί με μακροπρόθεσμα project για επενδύσεις ψηλού κινδύνου. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα κινηθούμε και πιο γρήγορα και θα εξασφαλίσουμε και τη βιωσιμότητα των επενδύσεων. Μακροπρόθεσμα. Τρίτον, θέλουμε να αφαιρέσουμε ε, τα εμπόδια που υπάρχουν στι επενδύσει του ιδιωτικού τομέα. Χρειαζόμαστε καλύτερο κανονιστικό πλαίσιο, χρειάζεται να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη για μια καινούρια Ευρώπη με μεταρρυθμίσει, διαφορετικέ μεταρρυθμίσει που θα δημιουργούν καλύτερο έδαφο, πιο γόνιμο έδαφο για τι επενδύσει. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ενιαία αγορά ε, στην ενέργεια, στους δημόσιους διαγωνισμούς, στις επιχειρήσεις, στις ε, ε, υπηρεσίες. Με αυτόν τον τρόπο θα αφαιρέσουν τα εμπόδια που υπάρχουν ε, για τις επενδύσεις. Επίσης, στον ψηφιακό τομέα το ίδιο. Υπάρχουν χώρες που έχουν ενιαία ψηφιακή αγορά. Στις ΗΠΑ είναι ένα παραδείγμα. Επίσης υπάρχουν πολλοί που θέλουν να επενδύσουν στον ενεργειακό τομέα, αλλά χωρίς ενεργειακή ένωση δεν μπορούν να το κάνουν. Θα πρέπει επίση να εμβαθύνουμε την ενιαία αγορά στου δημόσιου διαγωνισμού, στι κρατικέ προμήθειε δηλαδή και στι υπηρεσίε. Ε, θα με υποστηρίξουν η άλλη επιτροπή για την ολοκλήρωση τη ενιαία αγορά στι μεταφορέ, στον ψηφιακό τομέα και στην ενέργεια. Είμαι σίγουρο γι' αυτό. Θα συνεργαστώ επίση ε, με του ε, υπόλοιπου επιτρόπου για την ε, ενοποίηση τη ε, κεφαλαιογορά. Χρειάζεται αυτό για να στηρίξουμε και τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, ιδιαίτερω. Ε, η, τρίτη πλευρά της ενέας αγοράς, δηλαδή η τρίτη πλευρά του τριγώνου, είναι η πιο σημαντική για μένα στο έργο μας. Είναι πραγματικά η πλευρά του τριγώνου που θα αλλάξει την Ευρώπη για πάντα. Αυτό βέβαια δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Πρέπει όμως να αποφασιστικά να προχωρήσουμε μαζί. Είναι κοινή μας η ευθύνη. Κάθε μία από αυτές τις τρεις πλευρές του ε, τριγώνου είναι απαραίτητη για να προωθήσουμε τις ε, επενδύσεις. Κάθε μία από τι πλευρέ στηρίζει τις άλλε. Ε, κάποιοι λένε ότι τα χρήματα δεν είναι αρκετά. Δεν θέλουμε όμως να επιβαρύνουμε υπερβολικά τους ε, ε φορολογούμενους. Δεν χρειάζονται άπειρα χρήματα σε, στα ταμεία μιας τράπεζας. Χρειαζόμαστε λίγα χρήματα για να μοχλεύσουμε ε, πολύ περισσότερα και για να ξεμπλοκάρουμε επενδύσεις που ήδη είναι έτοιμες να γίνουν. Χρειαζόμαστε ένα μικρό ποσό για να αρχίσει να κινείται η μηχανή. Μετά η μηχανή θα λειτουργεί από μόνη της. Αν τα κρατημέλη θεωρούν ότι δεν είναι αρκετά αυτά τα κονδύλια, τις καλούμε να συνεισφέρουν και οι ίδιες και να, τα καλούμε να συνεισφέρουν και τα ίδια. Για να πετύχει το σχέδιο αυτό, τα κράτη-μέλη πρέπει να πάρουν ε, θαραλέες αποφάσεις και η ΕΤΕ πρέπει να παίξει το ρόλο της. Δεν έχουμε κάποια μαγική ράδο για να ε, μεταμορφώσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία. Είναι σημαντικό το σχέδιο αυτό. Αν υλοποιήσουμε και τα τρία στοιχεία του, θα αλλάξει για πάντα το επενδυτικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, ας δουλέψουμε όλοι μαζί για να ξαναφέρουμε τις επενδύσεις στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ως εκ τούτου ολοκληρώθηκε η συζήτηση.